Ε, από αύριο, 14 Οκτωβρίου, τρει μήνε στη διάθεσή μα για να τοποθετηθούμε. Βάσει του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 4, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα συνεδρίασε στις 10 Οκτωβρίου ε, και επικύρωσε τα διαπιστευτήρια και πρότεινε να κυρώσουμε τις εντολές του Αντρέα Ζινόιε με ισχύ από την 19η Ιουλίου 2011, Φιλίπ Ντεμπάκα από τις 7 Σεπτεμβρίου του 2011, Κάψουλου Στρούσοκ από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2011 και Μίκαελ Γκούσταυσον με ισχύ από την 22 Σεπτεμβρίου του 2011 ως εκ τούτου, σας προτείνω να επιβεβαιώσουμε και εμείς ε, την ισχύ των εντολών αυτών, των θητείων αυτών. Παρακαλώ, έχετε σχόλια. Δεν ε, βλέπω να ζητάει κανείς το λόγο, οπότε επικυρώνεται ε, και καλωσορίσατε.